Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Παρακαλώ πολύ να εγκαταλείψετε την αίθουσα ησύχω και με ταχύτητα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν το λόγο ε, με καλές συνθήκες το λόγο για την ε, συμπραγματική έκθεση του κυρίου Βέρνερ ε, Λάγκεν, ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Έχει το λόγο ο κύριος Μαούλου. Onorevole Maullo in aula. Κύριε Μαουλού, βρίσκεστε εντός της αιθούσης. La parola onorevole Mamikins. Επομένως, δίνω το λόγο στον κύριο Μαμίκινς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι η, ε, η οδηγία αυτή ε, για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την ε, ολοκλήρωση και την ε, υλοποίηση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών. Αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που εργάζονται και δραστηριοποιούνται εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξαρτήτως όμως της έδρας ε, των εταιριών αυτών ε, ή των δραστηριοτήτων τους, τα προϊόντα που διακινούν θα πρέπει να είναι απόλυτα υψηλής ποιότητας. Θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν ε, τη σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες για να επιλέγουν. Θα πρέπει όμως να ενθαρρύνεται και ο ελεύθερος ανταγωνισμός, ο απρόσκοπτος και χωρίς εμπόδια και θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εταιρείες αυτές η οδηγία που μας απασχολεί σήμερα θα μπορούσε να βοηθήσει για να μειωθεί και το κόστος των ασφαλίστρων. Γι' αυτό υπερψήφισα. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Χάναν. Κύριε Χάναν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Τώρα, αυτό που ε, ε, εννοούν μερικοί όταν, όταν μιλάνε για την ολοκλήρωση της κοινωνικής αγοράς, εννοούν ελευθερία ε, κινήσεων και αμοιβαία αναγνώριση υπηρεσιών όπως ε, έχουμε αμοιβαία αναγνώριση των ε, αγαθών. Αλλά εδώ όμως προαπαιτείται κοινή ρυθμιστική, κοινό ρυθμιστικό υπόβαθρο γιατί δεν σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετική νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών που όμως θα διαφέρει όσον αφορά ε, τους κανόνες από χώρα σε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι ορθώνονται ε, νέοι φραγμοί και επομένως ε, είναι ένα κακό στοιχείο της αγοράς εξ αρχής της οικοδόμησής της. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δημιουργούμε προσκόμματα στην ελεύθερη εγκατάσταση. Εμείς στο Ερεμένο Βασίλειο θέλουμε αυτή την ενιαία αγορά, αλλά δεν θέλουμε το κοινορθμιστικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άρνοτ. Η έκθεση αυτή ζητά αύξηση του επίπεδου προστασίας των καταναλωτών και φυσικά είμαι υπέρ. Αλλά το κάνει στο πλαίσιο της μείωσης της ανάγκης εθνικών μέτρων και περιορισμού της ικανότητας των εθνικών κυβερνήσεων να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις όπως το κρίνουν σκόπιμο. Επίσης περιορίζει ε, το πεδίο εφαρμογής ε, σε σχέση με τη μέχρι τώρα νομοθεσία και τις εξουσίες του ΕΙΟΠΑ. Πιστεύω ότι τέτοια μέτρα θα ληφθούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο παρά σε ευρωπαϊκό, σε κοινοτικό. Έχω και ένα άλλο πρόβλημα. Δίνουμε με την, με την οδηγία αυτή ε, αρμοδιότητα για κατεξοδότηση πράξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ουσιαστικά το δικαίωμα να νομοθετεί χωρί να περνάει από το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και τελικά η διορισμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει τι αποφάσει ε, για τα θέματα αυτά στο μέλλον, κάτι που είναι λάθο κατά τη γνώμη μου. Περνάμε στην έκθεση Ζουμπέρ, ο κύριο Ποσπίσιλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης ε, Ζουμπέρ γιατί θεωρώ ότι το θέμα της ε, παιδικής φτώχειας δυστυχώς βρίσκεται σε άνοδο και στην Ευρώπη. Κάτι που μας προβληματίζει. Πάνω από 1,6 εκατομμύρια, 8,6 εκατομμύρια παιδιών έχουν ε, πληγεί από την άνοδο αυτού του φαινομένου της παιδικής φτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Εγώ είμαι πολιτικός ε, της δεξιάς και είμαι υπέρ περιορισμένων δημοσιονομικών πολιτικών και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Πιστεύω όμως ότι τα μέτρα λιτότητας δεν θα πρέπει να πλήττουν τα παιδιά, να αυξάνεται η παιδική φτώχεια και να περιορίζεται η πρόσβασή τους στην παιδεία. Γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε στο μέλλον κοινωνικά ασθενείς γενναίες που θα δημιουργήσουν και προβλήματα στην εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Και αυτά δεν είναι κούφια λόγια. Διότι όταν δεν έχεις παιδιά δεν έχεις και μέλλον. Γι' αυτό κάθε πολιτική θα πρέπει να εκπονείται και να εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουμε στα παιδιά μας ποιοτική εκπαίδευση, πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, καθώς επίσης και συμπερίληψη ε, στην κοινωνική ζωή και όλα αυτά να είναι εγγυημένα. Δυστυχώς, παρά τα διαφορετικά και τα διάφορα σχέδια και προγράμματα που έχουμε, αυξάνεται και η φτώχεια και ο αποκλεισμό. Και μάλιστα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το φαινόμενο της φτώχειας από μόνο του είναι πάρα πολύ περίπλοκο, γι' αυτό θα πρέπει να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν καλύτερη πρόσβαση και στην μόρφωση και στη στέγη και στα ρούχα, στη σύντηση και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Εγώ πολύ ευχαρίστω υπερψήφισα την έκθεση και ευχαριστώ τον εισηγητή που την κατέθεσε. Ε, την εισηγήτρια μάλλον, γιατί η παιδική φτώχεια είναι σημαντικό φαινομένο. στα τέσσερα παιδιά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Απαράδεκτο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επενδύσουμε στην παιδεία, να αναχαιτήσουμε αυτό το φαινόμενο γιατί η παιδεία έχει σημαντικό ρόλο στη μείωση της παιδικής φτώχειας και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση των παιδιών στην παιδεία με ανάμειξη όμως ε, και των γονιών ε, και των ε, κυδεμόνων και επιτρόπων ώστε να πιστούν όλοι ότι η παιδεία είναι το εισιτήριο για να ξεφύγουν τα παιδιά από τη φτώχεια. Θα πρέπει να παιδίσουμε και σε θέματα στέγασης, σε προγράμματα υγιεινής διατροφής και στη δημόσια υγεία. Είμαστε ένα γυράσκον πληθυσμό. Γυράσκουμε λοιπόν, γι' αυτό και στο μέλλον θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο τα παιδιά μα, ε, τι νέε γενιές. Έχουμε και ηθικό καθήκον λοιπόν να παιδίσουμε από τώρα στα παιδιά, ε, γιατί από κάθε άποψη είναι ευνοϊκό και από κοινωνική και οικονομική. Ε, νομίζω ότι ο επόμενο ομιλητή δεν είναι στην αίθουσα και επομένω το λόγο έχει η κυρία Χουσμενόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Eurostat λέει ότι το ποσοστό των παιδιών σε παιδική φτώχεια από την Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία αγγίζει το 40%. Ταυτόχρονα έχουμε υποσυτισμό, εγκατάλειψη του σχολείου. Όλα αυτά είναι στοιχεία μιας ε, σίγουρης ε, πορείας κοινωνικού αποκλεισμού. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τα παιδιά στην ανάπτυξή τους να βοηθήσουμε του, τις μονογονεϊκές οικογένειες, ε, τους ε, άνεργους γονείς και γενικώ ε, τις μειονεκτούσες ομάδες. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε ώστε στα πλαίσια της θεπτικής του 2020 όλο και λιγότερα παιδιά να πλήττονται από το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον. ψήφισε υπέρ τη έκθεση, ε, ζητώντα δέσμευση από τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την παιδική φτώχεια και να περιορίσουν τι κοινωνικέ ανισότητε. Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεί σε ε, κατάσταση φτώχεια. 37% στη δική μου εκλογική περιφέρεια, κάτι που μας συγκλονίζει. Πολλοί ευρωβουλευτέ ε, τάχθηκαν υπέρ τη έκκληση ε, της έκθεσης ε, για ε, εγγύηση για τα παιδιά ώστε να έχουν όλα δωρεάν πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη, υγιεινή διατροφή και στην παιδεία και στις υπηρεσίες υγείας. Δεν θα πρέπει να περιορίζονται οι κοινωνικές δαπάνες και 640.000 επιπλέον παιδιά να περάσουν το κατόφλι της στόχης του χρόνου στο Λονδίνο. Ε, δυστυχώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται σε παιδική φτώχεια από το 2010 και θα συνεχίσουμε τη μάχη μας για να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο παντού. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Και εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή έστω και αν είχα κάποιες αμφιβολίες, ανεφέρθη ότι η τάση ε, είναι αυξητική όσον αφορά τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν τη φτώχεια. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό στήριξα αυτή την έκθεση. Ωστόσο πιστεύω ότι ε, το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους γονείς. Ε, είμαι ευτυχής γιατί ορισμένα στοιχεία που προέβλεπε η έκθεση δεν πέρασαν τελικά. Ας πούμε το ελάχιστο πρότυπο όσον αφορά την στέγαση των παιδιών. Πράγματι τα παιδιά πρέπει πρέπει να ζουν σε καλές συνθήκες, αλλά εάν οι γονείς δεν μπορούν να διασφαλίσουν ε, την, ε, μια τέτοια στέγη, ε, ποιος θα διασφαλίσει τη στέγη αυτή, το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οι εκκλήσεις ας πούμε που έχουν γίνει όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση δεν έχουν γίνει ακουστές στο Κοινοβούλιο, πώς μπορούμε να πιστέψουμε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή, λέει ο κύριος Κέλλη, γιατί θεωρώ ότι είναι ε, πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε τώρα για ε, μικρά παιδιά τα οποία ζουν σε συνθήκες ε, φτώχειας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται τα όσα πρέπει και τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση των Σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά γιατί δεν μπορούν ε, τα ίδια να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις είτε πρόκειται έλλειψη σε τροφή είτε πρόκειται σε στέγαση, σε εκπαίδευση κτλ. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα θέματα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ε, μία από τις πλουσιότερες περιοχές ε, του πλανήτη θα πρέπει να δείξει την διαφωνία της σε σχέση με αυτήν την παιδική φτώχεια θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Σόγκορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου και της Ευρώπης. Αντιμετωπίζουμε τεράστια πρόκληση το θέμα της εξάλληψης της παιδικής φτώχειας και στην Ουγγαρία δυστυχώς ε, αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς ε, ο αριθμός των υποσυτισμένων παιδιών και μάλιστα κάτι τέτοιο τον 21ο αιώνα. Θα πρέπει κατεπηγόντως ε, να βρούμε τα αίτια αυτής της φτώχειας ε, και να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτούς τους ε, στόχους και τις προκλήσεις και στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020 η εξάλληψη της παιδικής φτώχειας ε, και η εγκατάλειψη της σχολικής μόρφωσης θα πρέπει να είναι ύψιστες προτεραιότητές μας. Και με τη στρατηγική το 2020 θα πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος και της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, ε, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουν όλα τα κρατη το φαινόμενο αυτό, γιατί τα παιδιά που αναλαμβάνουν είναι το μέλλον της Υπήρου μας. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην ε, ιατρική φροντίδα και περίθαλψη, δικαίωμα στη στέγαση, ε, στην συμμετοχή ε, στις αποφάσεις που τους αφορούν. Όλα αυτά αναφέρονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, αλλά δεν καλύπτονται από πλευράς κυβερνήσεων. Μερικές κυβερνήσεις δείχνουν σαν να μην έχουν ακούσει ποτέ αυτές τις διατάξεις σε πολλό δε μάλλον ε, να τις εφαρμόσουν ένα στα τέσσερα παιδιά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούνται με φτώχεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το πιο πλούσιο μέρος του, του πλανήτη ε, και σε ορισμένες ε, χώρες της Ευρώπης η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να αλλάξει η ζωή των παιδιών. Αναφέρομαι σε μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία και την σωστή στέγαση. Η φτώχεια των ε, παιδιών ε, σημαίνει ε, γονείς σε συνθήκες φτώχειας, γονείς άνεργους. Ένα ρητό λέει ότι ο πολιτισμός προοδεύει όταν φυτεύουμε δέντρα που δεν θα χρειαστεί ποτέ να καθίσουμε κάτω από τη σκιά τους. Ευχαριστώ πολύ. Στην ε, δικιά μου γενιά είδαμε την μεγαλύτερη πτώση της ε, φτώχειας ε, σε ολόκληρη την ιστορία. Τα τελευταία 25 χρόνια όμως ε, η κατάσταση έχει ε, αλλάξει κυρίως στην Ασία και την ε, Αφρική. Βεβαίως η ένταξη των περιφερειακών αγορών σε μια παγκόσμια αγορά μπορεί να δώσει λύση στο, σε κάποιο, στο πρόβλημα αυτό της γενικής φτώχειας ας πούμε αγορά κινητών τηλεφώνων κτλ. Όλα αυτά τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρονται για την κοινωνική διάσταση του ε, προβλήματος και την αντιμετώπιση του μέσα από κοινωνικές ε, διαδικασίες ε, καθόλου δεν έχουν βελτιώσει την οικονομία. Πρέπει να σταματήσουμε την παρέμβαση, θα πρέπει να σταματήσουμε να νομοθετούμε και να βάζουμε πρότυπα. Είναι σημείο των καιρών στην έκθεση αυτή για ένα τόσο σημαντικό θέμα ανισότητας και παιδικής στόχιας και πάλι συζητούμε ένα θέμα για το οποίο κανονικά θα πρέπει να είναι ε, ε, υπεύθυνα τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις τους. Οι κρατικές αρχές και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι οι καλύτεροι ε, για να εντοπίσουν τι βελτιώσεις χρειάζονται και τι ανάγκες υπάρχουν και κάθε πολίτης να έχει ισότιμα, ίσα δικαιώματα. Δεν χρειάζεται η Ευρώπη να τα υπαγορεύει αυτά. Ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από την έκθεση. Ε, με ισορροπία θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή μας και θα μειώσουμε τις ανισότητες. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ε, κράτος και έθνος έχουμε αυτή την ευλογία να δίνουμε ε, κοινωνικά επιδόματα σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο στην κοινωνία για να έχουν μια μετάβαση στην αγορά εργασίας και να προστατεύονται οι πιο ευάλωτες ομάδες. Από την άλλη, ο στόχος και το κλειδί για να αυξηθεί η ισότητα στη ζωή για όλους είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η επιχειρηματική δραστηριότητα. Ευχαριστώ κύριο Σάρνοτ. Πιστεύουμε. Μπορεί να πιστεύουμε σε υψηλό επίπεδο ε, ε, υπηρεσιών και φόρων. Μπορεί να είστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση. Ε, μπορεί να είστε υπέρ της αναδιορμής του πλούτου και του εισοδήματος. Μπορεί να θεωρείτε ότι ε, γενικά επιδόματα καθολικά είναι καλύτερα από ε, στοχευμένα. Πολλοί πιστεύουν αυτά τα πράγματα, αλλά κατά την άποψή μου ε, είναι τελείως λάθος και ανομαλία να διαστρεβλώνεται αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα της παιδικής φτώχειας και να γίνεται αντικείμενο προώθησης και επιβολής αυτών των αριστερόστροφων πολιτικών. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ως χώρα είναι να αντιμετωπίσουμε την παιδική φτώχεια στο έδαφος μας. Το πρόβλημά μου με την έκθεση αυτή είναι ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα σε ε, θέματα ε, που είναι, και να τα βάλει στην έκθεση που είναι τόσο διαφορετικά από την παιδική φτώχεια και γι' αυτό καταψήφισα την επόμενη έκθεση για την πολιτική συνοχή και τι απελευθερωποιημένε κοινότητε και δίνω το λόγο στον κύριο Μαμίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική συνοχή δεν είναι απλώ ένα ακόμα μέσο και εργαλείο για να μπορέσουμε σταδιακά να μειώσουμε τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Βεβαίως μπορεί να γίνει και μέσω της πολιτικής συνοχής, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή πρέπει να δούμε και την κοινωνική περιφερειοποίηση και πώς αυτή μπορεί να αποφεύγεται. Γι' αυτό υποστηρίζω την έκθεση, είναι θετική ε, και θα μπορούσε να βοηθήσει για να λυθεί το πρόβλημα και να βγουν ορισμένες ομάδες και κοινότητες από το περιθώριο. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα αυτά, αλλά να αυξήσουμε και τη βιότητα συλλογής των στατιστικών δεδομένων και να καταλάβει όλος ο κόσμος ποια είναι τα προβλήματα, πόσο περίπλοκα είναι και πού βρίσκεται η αιτία του κακού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης ε, Ρέντκε που βελτιώθηκε από την αρχική της μορφή γιατί αρχικά ήταν πολύ γενική και κάλυπτε όλες ε, τις κοινότητες και τις θεωρούσε περιθωριοποιημένες. Τελικά ευτυχώς τροποποιήθηκε η έκθεση και έτσι μπόρεσα να την υπερψηφίσω. Η πολιτική συνοχής σημαίνει μείωση των ανισοτήτων και των αδικαιολόγητων διαφορών μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Πιστεύω ότι η πολιτική συνοχής είναι ταυτόχρονα και μια πολιτική που μας επιτρέπει να χτυπήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και μάλιστα, α, δυστυχώς, αυξάνεται ο αριθμός των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που είναι πολύ αρνητικό. Θα πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτές τις αρνητικές τάσεις. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ περιθωριοποιημένες κοινότητες ε, ε, χαρακτηρίζονται με βάση εθνικούς δείκτες από το κάθε κράτος μέλος. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μακροχρόνια ανεργία, η ελλειπής πρόσβαση στην παιδεία, ε, χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, αξιοπρεπεί συνθήκες στέγασης, πολιτικές διακρίσεων στις κοινωνικές υπηρεσίες υγειονομική περίθαλψης. Όλα αυτά είναι στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις, εταιρείες, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, ε, και να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης ε, και καλύτερη προσπάθεια ένταξης των περιθωριμένων κοινοτήτων και να μην υπογράφονται τέτοιες συμφωνίες εταιρικής σχέσης σε περίπτωση που συνεχίζεται αυτός ο αποκλεισμό. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των περιφερειών γιατί η παραμεθόριες κοινότητες είναι πιο ευεπίφορες στην περιθωριοποίηση εξαιτία της απομάκρυνσή τους, από το κέντρο. Χρειαζόμαστε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα που θα στηρίζουν και την επιχειρηματικότητα. Ο κύριος Χάναν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ξεκινούμε από σφαλμένη αρχή στην έκθεση αυτή. Η αρχή είναι ότι ο καλύτερο τρόπο για να μεταφέρουμε τι τις κοινότητε ε, στην κοινωνία είναι ο έλεγχο, ε, ο κυβερνητικό. Ε, όχι, δεν είναι αυτό το σωστό εργαλείο. Θα πρέπει να εθαρρύνουμε τους ενδιαφερομένου να αναλάβουν πρωτοβουλία και όχι να περιμένουν κοινωνικά επιδόματα, αλλά να επενδύσουν στις προσωπικές προσπάθειες. Ο καλύτερος τρόπος ένταξης είναι να βοηθήσουμε και να επιτρέψουμε το ελεύθερο εμπόριο και τι ε, συμβατικέ σχέσει χωρί κρατική παρέμβαση. Το καλύτερο σύστημα είναι αυτό τη ελεύθερη αγορά, όπω επισήμανε ο Μέλτον Φρίντμαν. Γιατί φέρνει σε επαφή ανθρώπου που μπορεί να μην είχαν καλέ σχέσει προηγουμένω. Νομίζω ότι το εξατομικευμένο σύστημα είναι το πιο αποτελεσματικό, γιατί θα είναι την συνέστηση και το να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Αυτό είναι πολύ καλύτερο από τα κοινωνικά κρατικά επιδόματα. Η έκθεση αυτή θέλει να εξασφαλίσει την πολιτική συνοχή να είναι προ όφελο των περιθωριομένων κοινοτήτων που είναι στο περιθώριο με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους. Στη Βόρεια Ιρλανδία τα διορθωτικά ταμεία σε διαδοχικές ε, προγραμματικές περιόδους ενίσχυσαν ε, θύματα της τρομοκρατίας με ε, η άρση των φραγμών που μπορεί να είναι φυσική, ψυχολογική και άλλη. Ε, και το κοινωνικό ε, ταμείο και άλλα ταμεία βοήθησαν ε, για να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η χρηματοδότηση και να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων. Σήμερα στη Βόρεια Ελλανδία, στην παρούσα προγραμματική περίοδο, η διαχειριστική αρχή έχει αγνοήσει τελείως τη συμμετοχή των γυναικών. Έχουν ε, βάλει εμπόδια και αυξήσει τα προβλήματα για τους δικαιούχους. Οι πολιτικές αυτές αγνοούν ε, τα ωφέλη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των άλλων ταμείων για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Έχει έρθει η ώρα ε, να τραβήξει καν αυτή η Υπουργού στη Βόρεια Ελλανδία, ο Αρμόδιος Επίτροπος Κάρβερ εγώ με χαρά λέω ότι είμαι απόγονος Ρωμά, ε, έχω τέτοια καταγωγή και χαίρομαι ε, για τη συμμετοχή μου σε ε, μια διάσκεψη στο Λονδίνο για θέματα Ρωμά. Η πολιτική μου θέση όμως δεν μου επιτρέπει να υποστηρίξω τη δράση που προτείνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά όλα πρέπει να λύνονται σε εθνικό επίπεδο και αυτό θέλει και η ομάδα μας και επιδιώκει. Αποχή ψήφισα, αλλά στο τέλος, αλλά στην αιτιολογική ε, σκέψη Q και στην τροπολογία 42 υπερψήφισα υπέρ των περιθωπημένων κοινοτήτων. Δεν με εκπλήσουν αυτά που λέει η έκθεση και η Βρετανική συντηρητική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε απαράδεκτα μέτρα που περιθωριοποιούν ακόμα περισσότερο τις κοινότητες αυτών των ομάδων και ε, μετακινουμένων πληθυσμών. Άρνοτ. Ε, ψήφισα αποχή ε, σε αυτή την έκθεση όπως και σε πολλές άλλες εκθέσεις. Τώρα, αν συμφωνώ ή όχι ότι ε, συχνά μεταχειριζόμαστε άσχημα ή έχουν κακή μεταχείριση οι μειονότητες, ναι, ε, έχουν, τους έχουν μεταγυριστεί με πέσιο τρόπο ορισμένες χώρες, ναι. Ε, πιστεύω ότι άραγε ότι οι χώρες ε, θα πρέπει κάτι να κάνουν έτσι ώστε να το θέμα αυτό, ναι φυσικά. Αλλά βλέπω και την έκθεση ε, η οποία προτείνει ενσωμάτωση, ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ωραία, να προσπαθήσουν οι συγκεκριμένες χώρες που έχουν αυτές τις κοινότητες να τις ενσωματώσουν. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν απήχα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην έκθεση ε, που αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Κάμπημαν είναι ο πρώτος. Κατεψήφισα αυτή την επικίνδυνη έκθεση, κύριε Πρόεδρε, γιατί... Ε, αποτελεί ακόμα μία προσπάθεια κατάλυσης της ε, εθνικής ανεξαρτησίας και ακερότητας μιας ε, χώρας. Εδώ ζητούμε και παραθέτω ε, τροποποίηση του Συμβουλίου Ασφαρίας η οποία θα δώσει μόνιμη θέση προσώπου στην Ευρωπαϊκή Έδρα, αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό όμως θα σήμαινε ότι ε, είναι το τέλος της δυνατότητας που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία, ε, να υποβάλει τις δικές της προτάσεις όσον αφορά ας πούμε την καταπολέμηση του φαινομένου του ISIS. Αυτή είναι μια επιθετική κίνηση στην οποία θα πρέπει να αντισταθούμε. Απ' την άλλη πλευρά είδαμε αυτό να συμβαίνει στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου όπου δεν έχουμε έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ασκήσουμε τη δικιά μας πολιτική. Άρα δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Ο κύριος Μαούλου δεν είναι εδώ. Ο κύριος Πασπισίλ. Ευχαριστώ. Εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης Βάρινεν, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εγκύψουμε στο θέμα της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με το σύνολο της οργάνωσης των του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεδομένη τη κατάσταση τη ασφάλεια στην Ευρώπη και τη επιδείνωση που έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, διαπιστώνουμε ότι τα διάφορα όργανα των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν άμεσα. Η σημερινή έκθεση δίνει όθηση στα κράτη-μέλη, ώστε όσα κράτη είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να ασκήσουν πίεση, ώστε να τροποποιηθεί το τρόπο λειτουργία του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά την νέα έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά σίγουρα η παρούσα κατάσταση είναι αρνητική. Και ελπίζω με την, με την σημερινή έκθεση να την βελτιώσουμε. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι ε, το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προβάλλεται ως κάτι σπουδαιότερο και μεγαλύτερο από ένα άθροισμα κρατών ή μια διακρατική ε, οργάνωση. Προσπαθεί να διευρύνει την επιρροή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλεται και προσπαθεί να τοποθετηθεί ε, ως ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές και οπαδός των ιδεών του ΟΗΕ. Παράδειγμα, καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, πολιτισμική ανταλλαγή και άλλα θέματα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πω ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν έλαμψαν πάντα δια της υποδειγματικής τους λειτουργίας από το τέλος ε, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ήταν πρωταγωνιστής παγκοσμίω οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ ενεργά και θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κλούν. Κύριε Πρόεδρε, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα Ηνωμένα Έθνη προϋποθέτει μία δομή που θα μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις παγκόσμιες ε, προκλήσεις και η συνθήκη της Λισαβόνας το αναγνωρίζει και επιτρέπει σε περίπτωση διεθνούς κρίσης ε, τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της είπα της εκπροσώπου για θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Στις στιγμές που μιλάμε αντιμετωπίζουμε τεράστιες παγκόσμιες προκλήσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνούμε ε, το ρόλο μας στα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να ασφαλίσουμε παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη, να συμβάλλουμε στην επίλυση των διαφορών, να προωθούμε θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα και να προωθούμε την οικονομική και οικονομική ανάπτυξη. Αυτή είναι η στόχη των Ηνωμένων Εθνών και εκεί θα είναι κέριος ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών. Το 1995, πριν από 60 χρόνια, προσχώρησε η Ιρλανδία στα Ηνωμένα Έθνη και χάρη σε αυτή τη συμμετοχή προωθήσαμε τους στόχους της εξωτερικής μας πολιτικής. Υπερψήφισα λοιπόν την έκθεση με ιδιαίτερη χαρά και θα συνεχίσω ευχαρίστω, θα συνεχίσω ευχαρίστω στη συμμετοχή μου στη συζήτηση για την αξιολόγηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Νέκοφ απουσιάζει, κυρία Σέιμουρ. Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας οργανισμός ε, που ε, εξηγεί όλα από μόνος του. Βέβαια η λέξη κλειδί είναι τα έθνη. Αν και κάποιοι θα θέλαν να είναι, ε, δεν ισχύει. Πρόκειται για μια ακόμη συνωμοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταλάβει έδρα στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έθνος και επομένω δεν έχει θέση στα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ υπερψήφισα την έκθεση και το έκανα πολύ ευχαριστώ. Μάλιστα είμαι σκέδος ηγητής του ΕΛΚ για την έκθεση αυτή και χαιρετίζω το γεγονός ότι ζητούμε καλύτερη συνεργασία και συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφορεί στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια στην ΟΕΕ. Έθνη. Οπότε ο ρόλο μα είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, είναι δύσκολη η σημερινή κατάσταση και μάλιστα βρισκόμαστε και εμεί στο στόχαστρο ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τι συνέβη στο Παρίσι, στι Βρυξέλλε. Οπότε Φαίνεται ότι θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα, να συντονιστούμε καλύτερα και μεταξύ μα, αλλά και με τα Ηνωμένα Έθνη, για να βοηθήσουμε τι ε, χώρε να αναπτυχθούν περισσότερο, για να εδρεωθεί η ειρήνη και να τεθεί ένα τέρμα στην τρομοκρατία. Η κυρία Μακοβέη δεν είναι στην αίθουσα, επομένω ε, θα δώσουμε τον λόγο στον επόμενο μιλητή, έχει Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σα σε αυτέ τι επεξηγήσει ψήφου. Συνεχίζουμε να ακούμε ότι ο ευρωφεντερελισμό έχει φτάσει στην κορυφωσή του και ότι τώρα υπάρχει όμω μια νέα πιο ευέλικτη προσέγγιση και έχουμε μια νέα επιτροπή που προσπαθεί να περάσει λιγότερη νομοθεσία και κατόπιν έχουμε αυτή τη συζήτηση που γυρνά μια έδρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι το, ο ανώτατος ορισμό του κρατισμού. Ε, η δική μου αντίρρηση ε, κοιτάξτε, φυσικά έχω αντίρρηση. Δεν περιμένω βέβαια να με καταλάβουν ε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αλλά εγώ θεωρώ ότι χτίζουμε εδώ ένα κράτος και μια κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει καμία έννοια ε, των ε, εθνών του ανήκει. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη ουσιαστικά το ίδιο συνέστημα ότι ανήκεις κάπου όπως στην Σουηδία, στην Πορτογαλία. Θεωρούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σημαία και να δημιουργήσουμε ένα κράτος πίσω από αυτό και να ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Δεν λειτουργεί. Ξέρετε ότι η ανθρωπίνη φύση είναι πιο ισχυρή από τα γραφειοκρατικά σχέδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αυτή τη συνεκτική ενότητα όπως έχουν τα κράτη. Ε, ευχαριστώ κύριε Άννα Ντότ, Λίτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε κάποια στιγμή στην αβεβαιότητας ε, και κατόπιν ε, των επιθέσεων στο Παρίσι. Είναι πολύ απογοητευτικό ότι αυτή η έκθεση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη επικεντρώνεται στην ένταξη και σε ένα σε μία και μόνη εντολή αντιπροσώπευσης για την Ευρώπη αντί να προωθήσει το συντενισμό και τη συνεργασία προς όφελος των πολιτών αντί να επιδιώκουμε έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη ε, να μιλάμε για το πόσο σημαντική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εντό των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να στρεψούμε την προσοχή μας όπως μπορεί η Ευρώπη να εκφράσει από κοινού τις εθνικές φωνές παρά να τις επισκιάζει. Εμείς πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση που εκλέγεται από τους πολίτες ε, της Βρετανίας και ένοπλες δυνάμεις μας ε, εκπροσωπούν καλύτερα ε, τη χώρα μας στο διεθνές επίπεδο. Δεν χρειαζόμαστε φωνή, χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία και συντονισμό και όπως ε, είπε και ο κύριος Κάμερον αυτή την εβδομάδα καλύτερη γνώση και συνειδητοποίηση για το πώς μπορούμε εθνικά να εργαστούμε σε καλύτερο επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Άρνοτ, παρακαλώ. Το ΟΗΕ είναι τα Ηνωμένα Έθνη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έθνος, δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι έθνος και δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έθνος. Ελπίζω να είναι σαφές λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να έχει ρόλο στον ΟΗΕ, στα Ηνωμένα Έθνη. Επόμενος παρακαλώ. James, η κυρία James. Κύριε Πρόεδρε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από τα κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εντός του ΟΗΕ και είναι μόνιμο μέλο. Η Γαλλία είναι το άλλο μόνιμο μέλο που έχει δικαίωμα βέτο. Δεν υποστηρίζω η αδίποτη προ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που υπονομεύει, υπονομεύει τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου σαν βασικό μέλο του ΟΗΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως να έχει κάποιες ε, ψευδεστήσεις μεγαλείου να αντικαταστήσει τα κράτη-μέλη σε αυτό το σώμα λήψη αποφάσεων αλλά εγώ ποτέ, ποτέ δεν θα υποστηρίξω το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γι' αυτό καταψήφισα όλα τα βασικά σημεία των ψηφοφοριών για το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τζέιμς. Etheridge. Ο κύριος Etheridge. Ευχαριστώ. Είναι πια πιο εύκολη επεξήγηση ψήφου θα δώσω ποτέ. UN. Είναι απλώ. Η Ηνωμένα Έθνη είναι ο ΙΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έθνο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα υπερήφανο κυρίαρχο κράτο και έθνο, Πάντα έτσι θα παραμείνει και ελπίζω ο Θεό να βοηθήσει ποτέ να μην βοηθήσω να αλλάξει αυτό. Πάντα θα καταψηφίσω τέτοια μέτρα και ελπίζω ο Θεό να μας βοηθήσει να κρατήσουμε την εξατησία μα την κυριαρχία μα και τη θέση μα την ξεχωριστή στον, ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή ήταν τελευταία επεξήγηση ψήφου για σήμερα. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση μέχρι τις 3.